Παρακαλώ καθίστε κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ για άλλη μια φορά να καθίσετε στις θέσεις σας. Άρχεται η συνεδρίαση της Ολομέλειας. Ξεκινούμε με την σημερινή μας ημέρα, τις εργασίες μας, με μια πανηγυρική επίσημη συνεδρίαση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να σας χαιρετήσω.